με τις ψηφοφορίες οι, τα πρακτικά θα υποβληθούν στην, στην ε, επόμενη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, καλό ταξίδι, λύεται η συνεδρίαση.